So, vielen Dank, meine Damen und Herren. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε και κύριοι. Okay, ich wäre dankbar, wenn die Damen und Herren. Θα σας παρακαλούσα κυρίες και κύριοι από τον τύπο να απομακρυνθείτε. Νομίζω πήρατε αρκετές φωτογραφίες. Okay. Νομίζω ότι καλό θα ήταν οι βουλευτές να μπορούν να βλέπουν τον Πρωθυπουργό όταν μιλάει. Σας ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα, λοιπόν, τα πρακτικά της χθεσινή συνεδρίασης, κύριε και κύριοι, είναι πλέον διαθέσιμα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν παρατηρήσει, σχόλια για τα πρακτικά αυτά. Αν όχι, θεωρούνται εγκεκριμένα τα πρακτικά. Αγαπητές κυρίες και κύριοι, σα παρακαλώ θα θέλαμε όλοι μαζί να χαιρετήσουμε τον κύριο Μιαλίτσκι στους, στα ε, θεωρία που είναι πρόεδρος των